της ε, Επιτροπής. Η κυρία Λουκασεύσκα έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, συζήτηση λοιπόν για την πρόοδο ε, της Σερβίας, την έκθεση πρόοδου για τη Σερβία. Παρακαλώ συνάδελφοι μπορείτε να βγείτε έξω. Έχει το λόγο το Συμβούλιο. Να υπογραμμίσω εδώ κάποια σημεία τα οποία περιλαμβάνονται και στο δικό σας ψήφισμα. Το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του καλωσορίζει την αρχή των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία στις 21 Ιανουαρίου του 2014 και τη διαδικασία ελέγχου από, αξιολόγηση συγγνώμη, από εκεί και πέρα. Η Σερβία έχει περάσει σε μια νέα φάση στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει μέχρι τώρα η σερβική κυβέρνηση. Είναι αφοσιωμένη στην προσπάθεια αυτή και αυτό έχει μεγάλη σημασία σε όλες τις, για όλες τις χώρες. Γιατί η μεταρρυθμιστική διαδικασία είναι πολλές φορές δύσκολη. Η Σερβία έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών και είναι προφανές ότι η προσπάθεια αυτή δείχνει και την αφοσίωσή τους. Νέοι στόχοι έχουν τεθεί στα πλαίσια του ανοίγματο νέων κεφαλαίων που απαιτούν και συγκεκριμένα προγράμματα δράσης. Έχει υπογραμμίσει θετικά το Συμβούλιο ότι τα κεφάλαια αυτά αντιμετωπίστηκαν ε, ενωρίς στα πλαίσια της διαδικασίας. Ο σεβασμός ε, των κανόνων του δικαίου είναι βασική προϋπόθεση και βρίσκεται στην καρδιά της διαδικασίας ένταξης, επηρεάζοντας όλους τους υπόλοιπους τομείς, οι οποίοι θα τεθούν στις διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει πρόοδος στα κεφάλαια αυτά, ε, παράλληλα με τις σύνολες διαπραγματεύσεις. Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έγινε το τελευταίο έτος και στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του δικαστικού σώματος, της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Σερβία συμμετέχει επίσης ενεργά και στα πλαίσια των περιφερειακών προσπαθειών επιβολής του νόμου. Αυτό είναι βασικό για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει τη Σερβία να εντατικοποιήσει λοιπόν τις μεταρρυθμιστικές της διαδικασίες. Συνεχείς προσπάθειες είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και να σημειωθεί πρόοδο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Η πρόθεση, η εφαρμογή και ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και σεβασμός των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα των Ρωμά, είναι βασικός στόχος. Η νομοθεσία, η νέα για την προστασία των μειονοτήτων πρέπει να εφαρμοστεί πλέον. Και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των μειονοτήτων. Πρέπει να δοθεί προσοχή και στην καταπολέμηση επίσης των διακρίσεων με βάση τις γενετήσιους προσανατολισμούς και τις θρησκευτικέ πεπιθήσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί επίσης η πλήρης ελευθερία έκφρασης. Υπογραμμίζουμε ταυτόχρονα την σημασία που έχει και η προστασία του περιβάλλοντος ελευθέρας εκφράσεως και ε, απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης. Ταυτόχρονα ε, πρέπει να βελτιωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και το πλαίσιο των ε, επενδύσεων. Πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω ε, μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει δημοσιονομική διασφάλιση, ανάπτυξη και απασχόληση. Προς την κατεύθυνση αυτή το Συμβούλιο συγχαίρει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενισχύει τους στόχους βελτίωσης της οικονομικής ε, ε, διακυβέρνησης. Είναι κάτι που θα στηρίξει ιδιαιτέρως τις προσπάθειες της Σερβίας να σεβαστεί και συνολικά τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Ένα βασικό τμήμα της διαδικασίας ενσωμάτωσης της Σερβίας είναι το πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας και οι καλές σχέσεις γειτονίας. Ως εκ τούτου λοιπόν καλωσορίζουμε τις συνεχείς ε, προσπάθειες της Σερβίας ε, ε, για τη βελτίωση των περιφερειακών μορφών συνεργασίας όπως η διαδικασία ε, συνεργασίας στο, στα νοτιοανατολικά της Ευρώπης και γενικά η βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η Σερβία θα πρέπει να συνεχίσει λοιπόν να εμπλέκεται θετικά και στην ε, προσπάθεια ε, ε, διαβουλεύσεων με το Κοσφοπέδιο. Έχουν υπάρξει αρκετές βελτιώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών και εδώ καλωσορίζω την επανέναρξη του διαλόγου υψηλού επίπεδου στις 9 Φεβρουαρίου και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το Κοσφοπέδιο για την δικαστική συνεργασία. Η εξομάλυνση των σχέσεων με την Πρίστινα ε, είναι ένας πολύ καλός στόχος. και συνδέεται θα έλεγα η προσπάθεια αυτή με ένα σημαντικό βήμα της προόδου της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις σερβικές προσπάθειες και την εφαρμογή ε, καλή την πίστη όλων των συμφωνιών στις οποίες καταλήξαμε μέχρι τώρα, έτσι ώστε το Κωσυφοπέδιο και η Σερβία να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή οδό και οι δύο χώρες, αποφεύγοντας η μία χώρα να δημιουργεί προβλήματα στην άλλη, εμπόδια στην άλλη. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν παράλληλη πρόοδος και παράλληλη πρόοδος και στις διαπραγματεύσεις συνολικά. Αγαπητά μέλη, το Συμβούλιο ζήτησε από τη Σερβία να συνεργαστεί και να ευθυγραμμιστεί και με την ΚΕΠΑ. Είναι βασικό ιδιαίτερα αυτή την εποχή για χώρες οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξουν ότι πιστεύουν στις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Τέλος, η Σερβία θα πρέπει να συνεχίσει να συνεργάζεται αποτελεσματικά με την Γιούλεξ και να συνεισφέρει σε μια ανεμπόδιστη εκτέλεση της εντολής της Γιούλεξ. Προσβλέπουμε λοιπόν στο άνοιγμα των επομένων κεφαλαίων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, now give the floor. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον Επίτροπο κ. Χάν. Ευχαριστώ, ναι, Πρόεδρε. Ξέρετε, κύριοι βουλευτέ, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον David Μακάλιστερ για το ψήφισμα ε, για την, προ, ε, την έκθεση πρόοδου για τη Σερβία του 2014. Είναι μια πολύ ισορροπημένη αξιολόγηση της πρόοδου της Σερβίας ε, και παρατίθεται τα ευρήματα από την έκθεση πρόοδου του 2014. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να βλέπουμε με θετικό πνεύμα της πρόοδου της Σερβίας και να προσβλέπουμε στο άνοιγμα των πρώτων κεφαλαίων. Οι διαπραγματεύσεις με τη Σερβία είναι σε εξέλιξη. Η χώρα έχει δεσμευθεί να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις και έχει καταφέρει πολλά στην εξομάλυση των σχέσεών της με το κοσυφοπέδιο. Αυτό αποτελεί και κλειδί για την σταθερότητα στην περιοχή. Η διαδικασία ελέγχου βαίνει βάση προγράμματος και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Είναι εντυπωσιακή η δέσμευση και ο επαγγελματισμός που δείχνει η Σερβία τους τελευταίους μήνες και αναμένεται ότι η πρόοδος θα συνεχιστεί και κατά τους επόμενους μήνες του έτους. Θα πρέπει η Σερβία να δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα για το κράτος δικαίου, για την εξομάλυνση των σχέσεών της με το κοσυχοπαίδιο, πράγμα το οποίο θα πρέπει ε, να αντιμετωπιστεί σύντομα στις αρχές της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το πλαίσιο διαπραγματεύσεων. Η ανάληψη των, του διαλόγου διαπραγματεύσεων πριν από ένα μήνα, μετά από διακοπή περίπου ενό έτου, ήταν κέρια σημασία. Η συμφωνία για το δικαστικό σώμα και για τη δικαιοσύνη γίνει στην Σερβία έχει ολοκληρωθεί και αυτό είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Ομάδες εργασίας θα εξετάσουν τώρα τα θέματα υλοποίησης και από τις δύο πλευρές και ελπίζω ότι θα έχουν σύντομα αποτελέσματα. Όταν θα αξιολογηθεί ότι έχει γίνει επαρκής πρόοδος θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο κεφάλαιο 35 και ελπίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει στο προσεχές μέλλον. Εξελίσσεται επίσης ε, σχετικό έργο όσον αφορά το κράτος δικαίου. Προσβλέπουμε στην υιοθέτηση προγραμμάτων δράσης που θα είναι αξιόπιστα και αποτελεσματικά και ελπίζω ότι αυτό θα συνεισφέρει στο άνοιγμα των κεφαλαίων 33 και 24 πριν από το τέλος του έτους. Η σερβική κυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα διακινδυνεύσει τα θέματα προόδου και δεν θα παρεμβαίνει στα θέματα του διαμεσολαβητού ούτε θα υπαναχωρεί στα θέματα της ελευθερίας έκφρασης. Η, έκφραση, η ελεύθερη έκφραση για τα μέσα ενημέρωσης ε, είναι ε, ένα θεμελιώδες ε, σημείο στο οποίο πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσει. Και τον, τονίζω μονίμω τον Πρωθυπουργό κ. Βούτση, με τον οποίο έχω τακτικέ επαφέ. εξετάζεται το κοινοτικό κεκτημένο και η ε, προσαρμογή στο κοινοτικό κεκτημένο και είναι σημαντικό να μην υπάρχουν διμερείς ε, ε, συγκρούσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο το συνολικό πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Σερβία στο δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μακάλιστερ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως μόνιμος ε, εισηγητής για τη Σερβία παρουσιάζω με τιμή του την έκθεση για την έκθεση πρόοδου. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γιαντράνκα Μισίμοβιτς, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της κυβέρνηση της Σερβίας που είναι παρούσα σήμερα. Θέλουμε με το να στείλουμε δύο μηνύματα Πρώτον, η Σερβία είναι καθοδόν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 ήταν μια σημαντική χρονιά για την Σερβία που η επίσημη, η επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων έγινε στις 21 Ιανουαρίου. Είμαι πεπισμένος ότι ο Πρωθυπουργός κ. Βούτσιτς και η κυβέρνησή του έδειξαν δέσμευση υπέρ της ενοποίησης, αντιμετώπισαν ξεκάθαρα τις αναγκαίες ε, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, κάτι που αξίζει την υποστήριξή μας. Τους πρόσφατους μήνες το Κοινοβούλιο της Σερβίας υιοθέτησε μια σειρά σημαντικής ε, νομοθεσίας για τα, για τα μέσα ενημέρωσης, την ιδιωτικοποίηση, την ε, πληροφο... τους, τους φορολογικούς πληροφοριοδότες κλπ. Ωστόσο, μια πλήρης ε, υλοποίηση των πολιτικών αυτών είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ενταξιακή προοπτική. Δεύτερον, κλειδί στις διαπραγματεύσεις είναι οι βασικές ε, οι βασικές αλλαγές μεταξύ των οποίων κράτο δικαίου, οικονομική διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση της διοίκηση, προσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας με την ευρωπαϊκή και εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσμοπέδιο πόσο καιρό θα κρατήσουν οι ενταξιακές διαχρηματεύσεις. Αυτό εξαρτάται κατά βάση από τη βούληση και την ικανότητα της Ρωσία να αντιμετωπίσει και να υλοποιήσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είμαι ωστόσο πεπισμένος ότι η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί. Το τρένο του Βελιγραδίου είναι στο δρόμο για τις Βρυξέλλες. Ας παροτρύνουμε την Σερβία να μείνει στην ευρωπαϊκή γραμμή. Και θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την καρποφόρα συνεργασία που είχαμε. Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε ένα ρεαλιστικό, δίκαιο και ισορροπημένο κείμενο, κάτι που νομίζω ότι πετύχαμε. Ευχαριστώ. Επόμενος αγωγητής, η κυρία Φαγιόν, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε, συνάδελφοι, επίτροπε. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη κάθε φορά που βλέπω μπροστά μου ένα κείμενο που περνάει ένα θετικό μήνυμα και που εμπνέει αισιοδοξία. Ευχαριστώ τον εισηγητή David ε, για που παρουσιάζει την πρόοδο της Σερβίας υπογραμμίζω τη σημασία των βημάτων που έχουν γίνει μέχρι τώρα και είμαι αισιόδοξη για το μέλλον. Ταυτόχρονα ωστόσο εκφράζω την ανησυχία μου όταν βλέπω τάσεις και πιέσεις που διαπιστώνονται τον τελευταίο καιρό για θέματα που έχουν να κάνουν μόνο με διμερείς σχέσεις με την Σερβία. Νομίζω ότι όταν ζητούμε από την Σερβία να επανεξετάσει την ομοθεσία της για τα εγκλήματα πολέμου, δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι στην έκθεση η οικουμενική δικαιοδοσία στα θέματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου είναι κάτι που επιβεβαιώνεται από την διεθνή νομολογία. Οι χώρες της Ευρώπης έχουν αντίστοιχη νομοθεσία. Η Επιτροπή έχει την ίδια άποψη, ενώ επιπλέον η φυστάμενη νομοθεσία είναι πιο αποτελεσματική και επιτρέπει την δίκη ούτως ή άλλως και απουσία της πιθανής εθνικής νομοθεσίας. Ζητώ λοιπόν να καταψηφίσετε την τροπολογία υπαριθμών 3. Να θυμίσω επίσης ότι συζητήσαμε το ψήφισμα ένα ψήφισμα με αντίστοιχο σκεπτικό που δεν ήταν αποτελεσματικό. Την ίδια, εκείνη τη φορά είχα τονίσει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε το κοινοβούλιο για να κάνουμε εθνικές πολιτικές. Η Σερβία έχει τεράστια ευθύνη στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, έλαβε την ευθύνη να βελτιώσει τη σχέση της με την περιφέρεια. Μην ξεχνάμε τη συμφωνία αρχής για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Κωσυφοπέδιο. Ζητώ να γίνουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό και θα είμαι στο Βελιγράδι σύντομα. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδίω την ε, εξομάλυνση των σχέσεων με το κοσφοπέδιο. Κυρία Φαγιόν, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Κυρία Πίτερ, έχετε... Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Φαγιόν, ότι δεν ξέρετε από ό,τι φαίνεται ότι αυτά που αναφέρατε εφαρμόζονται και για τους δικούς σας πολίτες, όχι μόνο για τη Σερβία. Συνεχίζετε λοιπόν να έχετε την άποψη ότι ο νόμος αυτός δεν παραβιάζει τη διεθνή νομοθεσία. Κάποιος που συλλαμβάνεται και δικάζεται βάσει του νόμου αυτού, πώς θα ε, αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Την περίμενα την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, περίμενα την ερώτησή σας για τα εγκλήματα πολέμου, για τη Σερβία. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει, νομίζω, με ε, πολύ καλό τρόπο τις συνθήκες στα πλαίσια των οποίων θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις γύρω από τα κεφάλαια 23 και 24. Η αλλαγή του νόμου στη Σερβία λοιπόν στο συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε ό,τι έχει σχέση με την διασενοριακή δικαιοδοσία είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει σε μία χώρα φυσικά αλλά σε περισσότερες. Περνάμε στον επόμενο ομιλητή Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εκπρόσωπε της Προεδρίας, κύριε Μακάλιστερ, η εκθεσή σας είναι μια σωστή έκθεση είναι μια έκθεση η οποία δικατοπτρίζει με αντικειμενικό τρόπο τις εξελίξεις στη χώρα αυτή. Έχει υπάρξει πρόοδος, υπάρχει ετοιμότητα για διάλογο, υπάρχουν όμως και προβλήματα. Όχι μόνο εσωτερικά προβλήματα όπως το θέμα της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας των ΜΜΕ. Υπάρχουν θέματα ε, και σε ε, σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, υπάρχουν θέματα με την Κροατία, Κάποιοι νόμοι οι οποίοι υιοθετήθηκαν δεν εφαρμόζονται στην ουσία. Σαν παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής ε, ε, μαθημάτων στη βουλγαρική γλώσσα. Αυτά όλα πρέπει να τεθούν και πρέπει η Σερβία να τα λύσει εφόσον θέλει να ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο. Βάγκλ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος λοιπόν και της ομάδας των φιλελευθέρων υποστηρίζω το συγκεκριμένο ψήφισμα και την προσπάθεια την ιδιαίτερως επικοδομητική την οποία έχουν κάνει μέχρι τώρα ε, οι εισηγητές και συγκεκριμένο ο κ. Τα επιχειρήματά του είναι ιδιαίτερως πιστικά και μπορούμε να αξιολογήσουμε θετικά τις σερβικές προσπάθειες. Είναι προφανής η πρόοδος την οποία έχει επιτελέσει η συγκεκριμένη χώρα οι μεταρρυθμιστικές διαδικασίες ήσαν αποτελεσματικές και η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Το ψήφισμα υπογραμμίζει αρκετούς τομείς τους οποίους θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω προσπάθειες όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η σταθεροποίηση της νομοθεσίας, η νομική ασφάλεια στον τομέα της επιχειρηματικότητας και φυσικά ο σεβασμός των μειονοτήτων κάθε είδους κτλ. Η Σερβία λοιπόν είναι μια σημαντική χώρα και σημαντικός παράγων περιφερειακής σταθερότητας. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ράνσβορτ, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω ότι η Σερβία είναι βασικός πυλώνας των Βαλκανίων και χωρίς σταθεροποίηση της Σερβίας δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τις χώρες των Βαλκανίων. Θέλω να τονίσω ότι η χώρα αυτή χρειάζεται μακροοικονομική βοήθεια διότι έχει το μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων. 700.000 πρόσφυγες. Επίσης ε, με τις πλημμύρες ε, ε, πλημμύρισαν και ορυχεία άνθρακα και ε, άλλος ένας λόγος να βοηθήσουμε τη Σερβία να δημιουργήσει υποδομές στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουν γίνει βεβαίως πρόοδοι στα θέματα υδροηλεκτρικών σταθμών ενέργειας, αλλά παραμένουν κάποιες επιφυλάξεις γιατί ο τομέας, ε, και πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε κάτι γιατί ο τομέας της ενέργειας είναι σημαντικός και για τις γειτονικές χώρες. Αναγνωρίζουμε την, ε, τις μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει ακόμη να γίνουν ε, προσπάθειες στον τομέα του κράτους δικαίου, της καταπολέμησης, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μια χώρα που αξίζει την προσοχή μας και είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να χρησιμοποιήσει το δυναμικό που έχει και που είναι δυναμικό για όλη την περιφέρεια. Ο κύριος Σόλτες είναι ο επόμενος μιλητής για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μακάλιστερ για την εξαιρετική έκθεσή του για την πρόοδο της Σερβίας και τον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και για το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε σε όλες τις συμβιβαστικές λύσεις και για τις εξαιρετικές συζητήσεις που είχαμε. Το έγγραφο του κ. Μακάλη είναι εξαιρετικό και θα το υποστηρίξω. Η Σερβία έχει κάνει πολλά σημαντικά βήματα έχει ξεκινήσει πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις και θα πρέπει ε, να τονίσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, στη Σερβία και στον δικαστικό τομέα. Αναζητούμε μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για το κράτος δικαίου. Η διαφθορά είναι ένα σημαντικό θέμα στην Σερβία και η σχετική διαδικασία έχει δρομολογηθεί. Θα χρειαστεί όμως ακόμη χρόνος. Είμαι πεπισμένος ότι η Σερβία θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές και ότι θα προσπαθήσει να επιτύχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βλέπω ότι η Επιτροπή έχει δουλέψει αποτελεσματικά όσον αφορά την διαφάνεια γιατί είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να ελέγχουμε τη διαφάνεια στην χρησιμοποίηση δημοσίων κονδυλίων και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου βλέπουμε ότι υφίσταται πραγματικές προσπάθειες. Υπάρχει ανεργία στη Σερβία, υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης των μέσων ενημέρωσης και αυτό είναι ένα θέμα που πολύ συχνά αναφέρεται και λαμβάνω και πολλά μηνύματα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για το θέμα αυτό. Πάντως είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Για ένα λεπτό ο κύριος Κάβερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η νεοϊπερελιστική επέκταση της Σερβίας στην, ε, της Ένωσης στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβία μας έκανε να χάσουμε την ε, γενικότερη εικόνα της σχέσης Σερβίας και Ρωσίας. Ξεχνάτε τους στενούς πολιτιστικούς δεσμούς που έχει η Σερβία με τη Ρωσία μέσω της κοινή ορθόδοξης παράδοσης. Η Σερβία γίνεται ένα ακόμα πιόνι στον αγώνα, μας, στον αγώνα της Ρωσίας εναντίον σας. Αν είχατε σεβασμό για το, λαό της Σερβίας θα καταλαβαίνατε ότι ε, αυτό που θα είναι σημαντικό είναι η συμφιλίωση και η συνεργασία. Αντί να κάνουμε τη Σερβία ένα άλλο υποτελεί τη επιτροπή θα πρέπει να αφήσουμε την Σερβία να γίνει ένα σημαντικός διαμεσολαβητή μεταξύ Ευρώπης και Ρωσία σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για την ασφάλεια τη Ανατολική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα κύριε Κάρβελ. Παρακαλώ. Ε, η Ρουμανία είναι και αυτή η ορθόδοξη χώρα θα πρέπει και εμείς να έχουμε την ίδια στάση έναντι της Ρωσίας, να δεχθούμε δηλαδή μια ειδική σχέση και να... με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι εκτιμούμε τις ευαισθησίες της κατάστασης ό,τι αφορά τις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Είναι μια καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε τη Σερβία ως διαμεσολαβητή αν αν εντάξουμε τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζετε το παιχνίδι του κυρίου Πούτιν και τον κάνετε ακόμα πιο επιθετικό. Ευχαριστώ. Κύριε Μουρβάη. Ευχαριστώ. Η έκθεση για την Σερβία θα ήταν αξιόπιστη αν υπήρχε ένας κατάλογος μεταξύ των οποίων τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα του ανθρώπου που θα έπρεπε να τηρεί μετά από έτοιμά μας η Σερβία για ιστορικές, εθνοτικές μειονότητες. Για παράδειγμα τους 300.000 Ούγγρους στην καταγωγή στην Βοηβοδίνα. Αλλιώς δεν θα μπορεί να ενταχθεί η Σερβία στην Ένωση. Η Σερβία κατά την άποψή μας θα έπρεπε να δώσει πλήρη ε, αυτοδιοίκηση και δικαίωμα αυτοδιάθεση στην περιοχή της Βοηβοδίνας βάσει και του μοντέλου του Νοτιού Τυρόλου. Η... Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή στην ε, Βοηβοδίνα καταργούνται τα ιδιωτική αδιοφωνική σταθμή θα έπρεπε η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, ισότητας των δικαιωμάτων των Ούγγρων στη Βοηβοδίνα. Ο κύριος Κούκαν. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι ε, έχουν θέσει μπλε κάρτα, αλλά είσαστε στον κατάλογο ομιλητών. Θα δώσω μπλε κάρτα μόνο σε όσους δεν είναι ομιλητές. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σερβία καταβάλει πρόοδο στην ενταξιακή της προοπτική και ελπίζω η ισορροπημένη έκθεση και, το, και η ισορροπημένη έκθεση του κ. Μακάριστερ το αναγνωρίζει αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξει δέσμευση στο πλαίσιο αυτό σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και να ενισχύσει τη δουλειά της κυβέρνησης στο θέμα αυτό. Ζητούμε να ξεκινήσουν και σωστά οι διαπραγματευτικά κεφάλαια θα είναι κρίσιμο να μπορέσει η Σερβία να προχωρήσει τις, ε, τη διαδικασία μεταρρύθμισης. Υπήρξαν δύσκολες μεταρρυθμίσεις, περιμένουμε συνεχή πρόοδο στην ε, μεταρρύθμιση των, της δικαστικής αρχής. Υπογραμμίζω στο σημείο αυτό την ανεξαρτησία κάποιων οργάνων όπως του συνήγορου του πολίτη, αλλά και θεμάτων που σχετίζονται με τις πιθανότητες καταχρήσεως ε, θέσεις. Η Σερβία πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο με το κοσφοπέδιο. Η ιδέα υποστήριξη από την πολιτική ελίτ και την κυβέρνηση στη διαδικασία αυτή είναι κλειδί για τη σταθερότητα της περιοχής. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Ο κύριος Φρουντζουλίτσα. Η Ρουμανία είναι γειτονική χώρα προς τη Σερβία και έχουμε και μακρά παράδοση φιλίας με τη χώρα αυτή. Υποστηρίζουμε μια προοπτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την Σερβία, αλλά για όλες τις πρώην γιουκοσλαβικές δημοκρατίες και για την Αλβανία και για τη Μολδαβία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Σερβία έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Χρειάζονται πολλές βελτιώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, ε, την διαφάνεια στη χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, τη διαφθορά. Πιστεύω ότι στις διαπραγματεύσεις μας με όλες τις υποψήφιες χώρες θα πρέπει να έχουμε κατά νου ξεκάθαρα τις ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες. Ο στόχος της επίτευξης σταθερότητας στην περιοχή είναι πολύ σημαντικός αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις βασικές ελευθερίες στα Βαλκάνια. Υποστηρίζω τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Διεύρυνσης στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα όμως θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρα πολιτική θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ένα λεπτό, ο κύριος Ουγιασδόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την ε, ειλικρινή έκθεση που είναι ταυτόχρονα και αισιόδοξη. Καταγράφει την πρόοδο της Σερβίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Χάρηκα όταν η Σλοβενία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Κροατία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω ότι θα δείξουμε καλή θέληση και θα ανοίξουμε την πόρτα και στη Σερβία. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μιλά με μία φωνή στα θέματα αυτά. Θέλω να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Βρετανός συνάδελφος από το κόμμα του κυρίου Φαράζ. Υπάρχει μία διάμεση ζώνη μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης. Αν δεν ανοίξουμε εμείς την πόρτα στη Σερβία, αν εμείς δεν τους δείξουμε καλή θέληση, θα μπουν στη ζώνη επιρροής της Ρωσίας. Και δυστυχώς το κόμμα του κυρίου Φαράζ μίλησε με τη φωνή της Μόσχας για άλλη μια φορά. Εμείς πρέπει να μιλάμε με τη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο κύριος Γιάκοβιτς είναι ο επόμενος ομιλητής. Συγχαίρουμε λοιπόν την κυβέρνηση της Σερβίας που συνεχίζει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Είναι κάτι το οποίο θα συνεισφέρει στη σταθερότητα του συνόλου των Βαλκανίων. Ο βέλος της Σερβίας πάντα ήταν σημαντικό στα Βαλκάνια. Και οι τελευταίες εξελίξεις σε χώρες ε, όπως η Σερβία και η Αλβανία είναι θετικά μηνύματα. Εφόσον η Σερβία συνεχίσει στην πορεία αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να την αποδεχθούμε ως μέλος το ταχύτερο δυνατόν. Πρέπει να συνεχιστούν βέβαια οι μεταρρυθμίσεις. Είναι σωστό το πρόγραμμα της κυβέρνησης και θα πρέπει να δούμε και την δυνατότητα την οποία έχει η Σερβία, παρουσιάζει η Σερβία στον τομέα της ενέργειας. Θα πρέπει ίσως να συμπεριληφθεί και στο πρόγραμμα των στρατηγικών επενδύσεων του κ. Γιούνκερ. Πλένκοβιτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Εισηγητή, σας ευχαριστώ για μια πολύ καλή έκθεση για τη Σερβία. Είναι ένα πολύ καλό κίνητρο για την κυβέρνηση της χώρας αυτής για να συνεχίσει την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει σωστή αναφορά στις μειονότητες και στον σεβασμό των συμπεφωνημένων και σε επιμέρους θέματα όπως το θέμα των, ε, ε, των προσώπων τα οποία έχουν εξαφανιστεί και αναζητούνται, των αγνοουμένων. Υπήθεται και το θέμα εδώ της ε, διασυνοριακής επίσης δικαιοδοσίας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να τεθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο θα παρουσίαζε και μια κάποια πρωτοτυπία. Ε, καλά έκανε η Επιτροπή και έθεσε το θέμα διότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια νομική αβεβαιότητα σε Ευρωπαίους πολίτες όπως ε, και εννοώ τους Κροάτες πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμίσει το δικαστικό της σύστημα η Σερβία. Έχω δύο μπλε κάρτες, αλλά ε, έχουμε καθυστερήσει και θα δεχθούμε μία. Μία λοιπόν από την κυρία Τσβίτσκα. Ευχαριστώ. Κυρία Πλένκοβιτς, αναφερθήκατε το θέμα της ε, δικαιοδοσίας ε, για τελεστέντα δικήματα πιθανώς σε άλλες χώρες. Ίσως εδώ να υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως να μην το καταλαβαίνετε κι εσείς και η κυρία Φαγιόν. Πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι εννοούμε εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να σταματήσουμε τη Σερβία. Θέλουμε να τη βοηθήσουμε στην πορεία της προς την Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν περάσει κάποιοι μήνες από τότε που τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά στην ε, Αρμόδια Επιτροπή. Ελπίζω να μην προσθέσαμε στη σύγχυση που πιθανώς μπορεί να υπάρχει. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά τα κατανοούν οι συνάδελφοι Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες υιοθετούν την αντίληψη αυτή. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με μία χώρα, αλλά έχει να κάνει με τις πιθανότητες δίωξης για εγκλήματα πολέμου. Προφανώς είμαστε κατά της ασυλίας και της ατιμορρησίας. Από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να δημιουργείται νομική αβεβαιότητα ε, για τους ε, Κροάτες ε, πολίτες. Να σας θυμίσω ότι στις μπλε κάρτες ερωτήσεις τίθενται, όχι δηλώσεις. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των αγωγητών. Ο κύριος Τσάνι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πλένκοβιτς. Πρόκειται για μια θετική έκθεση που καλύπτει όλους τους τομείς πρόοδου της σερβικής κυβέρνησης αλλά και τους τομείς εκείνους, τα πράγματα που περιμένουμε ακόμα από την Σερβία. Επίτροπε, θέλω να τονίσω δύο πράγματα. Πρώτον, οι υποψήφιες χώρες πριν την ένταξη πρέπει να συμμορφωθούν με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Αναμένουμε να συμφωνήσει η Σερβία επιβάλλοντας τις κυρώσεις κατά της ε, Ρωσίας. Η Ουγγαρία είναι πολυεθνική χώρα. Εμείς είμαστε πολυεθνική χώρα και αυτή είναι πολυεθνική χώρα. Αυτό σημαίνει σεβασμό των εθνικών μειονοτήτων, κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπανέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόοδο που πέτυχε η Σερβία στην Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης. Επίσης, την δέσμευση της σερβικής κυβέρνησης υπέρ της ευρωπαϊκής εντοποίησης. Η νομοθεσία που υιοθετείται ωστόσο πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε επίπεδο. Εφιστώ λοιπόν την προσοχή σας στην ανάγκη υλοποίηση της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, την πρόσβαση στον τύπο και την λατρεία όλων των θρησκειών στις χώρες αυτές αλλά και την εκπροσώπηση των μειονοτήτων σε κάθε επίπεδο τοπικό και περιφερειακό και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει ένα εθνικό πρόγραμμα για τις εθνικές μειονότητες στις συζητήσεις ε, του κεφαλαίου 23. Η ένταξη της ε, Σερβίας θα συμβάλλει για τη σταθερότητα και για τον σερβικό πληθυσμό αλλά και για την Ευρώπη θα δώσει και η καλύτερη διαχείριση των εθνικών μειονοτήτων θα ενισχύσει την διαδικασία ένταξης. Συγχαίρω τον κύριο Μακάλιστερ, είχε μια πολύ σωστή και ισορροπημένη προσέγγιση στο κείμενό του. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για τις χώρες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να τονίζουμε ότι οι χώρες θα πρέπει να επιλέγουν μεταξύ φιλελεύθερης δημοκρατίας και αυθαίρετων ε, αυταρχικών καθεστώτων. Υπάρχουν υποχρεώσεις που βασίζονται στις δημοκρατικές αρχές και υπάρχουν τα άλλα συστήματα τα οποία καταστρέφουν την ειρήνη τη Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Δεν μπορεί να επιλέξει κανείς πάνω από ένα σύστημα. Η Σερβία ακόμη θέτει πολλά ερωτήματα ε, για το σημείο στο οποίο βρίσκεται οι πράξεις σε σχέση με τη Ρωσία αποτελούν δήλωση. Αυτή τη στιγμή οι χώρες της Ανατολικής Συμμαχίας όπως η Ουκρανία θα, ε, ε, να είναι, ε, φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι άλλες χώρες που φαίνονται στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό τονίζω προς τη Σερβία ότι δεν είναι δυνατόν να έχει και τα δύο ταυτόχρονα. Ένα λεπτό, κύριος Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο η Σερβία ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις και έδειξε προθυμία να ακολουθήσει την οδό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τώρα αυτή η προθυμία θα πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη. Η Σερβία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υποχωρήσει σε πίεση από τρίτες χώρες. Γι' αυτό Επίτροπε, θα πρέπει να βοηθήσουμε τη Σερβία. Η Σερβία έχει, σωστές, έχει ακολουθήσει σωστές πολιτικές όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όχι πάντοτε όμως. Η βουλγαρική μειονότητα συνεχίζει να έχει προβλήματα όσον αφορά την εκπαίδευση στην μητρική τους γλώσσα. Υπάρχουν κάποιες προφάσεις ε, που προβάλλονται για, το, για τη μη μετάφραση των σχολικών κειμένων ε, στα βουλγαρικά. Θα πρέπει η Σερβία να συμφιλειωθεί με την ιστορία της ε, και να ανοίξει ε, τους φακέλους των μυστικών και ειδικών υπηρεσιών και να δώσει τα αρχεία στις πρώην ε, Ιουκοσλαβικές δημοκρατίες. Είναι σημαντικό η πολιτική ολοκλήρωση να συμπεριλαμβάνει και τις συνοριακές περιοχές όπου ζουν πολλές μειονότητες και η κατάσταση είναι πολύ φτωχή. Κύριε Θεοχάρους. Υποστηρίζουμε στεναρά την ένταξη της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχαίρω τον κύριο Μακάλιστερ για την εξαίρετη έκθεση που έχει ετοιμάσει. Πιστεύω ότι η χώρα αυτή και ο σερβικός λαός χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά στο θέμα της ανάπτυξης των δημοκρατικών θεσμών και των μεταρρυθμίσεων. Η Σερβία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει προς αυτή την ε, κατεύθυνση. επιπλέον έχει δύο βασικά πλεονεκτήματα το ένα είναι ότι μπορεί να καταστεί ένας σταθεροποιητικός παράγοντας στα βαλκάνια και το άλλο ότι έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος μπορεί να ξαναγίνει ένα βιομηχανικό και αγροτικό κέντρο στην περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των σχέσεων με την Ρωσία, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε για μεν την Τουρκία να μην βλέπουμε ότι ούτε την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ακολουθεί έχει άριστε σχέσει με τη ρωσία και δεν οφείλεται αυτό στην ορθοδοξία η μια είναι μουσουλμανική η άλλη είναι ορθόδοξη και για τη σερβία αυτό να αποτελεί ε, αρνητικό στοιχείο. μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα συνεννόηση με την ρωσία. η σερβία έχει επιδείξει εξαιρετική συνεργασία με το ειδικό διεθνέ δικαστήριο για τα εγκλήματα πολέμου στην πρώην γιουγκοσλαβία αλλά και για το ζήτημα των διαφορών με το κωσυφοπαίδιο μια περιοχή που συνιστά την κοιτίδα για τους Σέρβους του σερβικού πολιτισμού. Έχω κι άλλα να πω, αλλά ευχαριστώ αφού δεν έχω χρόνο. Thank you. For one minute, Mr. Daly, please. Ένα λεπτό, κύριος Daly. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπαμε πολλά για την έκθεση για τη Σερβία. Είπαμε ότι είναι μια ισορροπημένη έκθεση και χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ τον κύριο Μακάλιστερ για την πολύ ισορροπημένη αυτή η έκθεσή του. Μιλήσαμε για τα σωστά βήματα της σερβικής κυβέρνησης καθώς και για τις προκλήσεις που παραμένουν. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη σερβική κυβέρνηση στο δρόμο της προς την ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ουγγαρία είναι μια γειτονική προ τη Σερβία χώρα και έχει ένομο συμφέρον ε, στο να είναι η Σερβία μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική πολιτική και στην οικονομική πολιτική και στι καλές, ε, ε, στις σχέσεις καλής γειτονίας που έχουν μεγάλη σημασία. Είναι προ όφελο της Ευρώπης να βοηθήσει και την εθνική και τους Ούγγρους της Σερβίας, την εθνική αυτή μειονότητα και τα δικαιώματά της. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή της Βοηβοντίνα, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον των ε, Ούγγρων στην Σερβία. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα δεχθώ μπλε κάρτες. Ε, κυρία Μορβά, έχετε ήδη λάβει το λόγο. Θα ε, δεχθώ τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye, ένα από κάθε ομάδα. Κύριος Μπόγκοβιτς, ένα λεπτό. Εγώ Δέχομαι τις προτάσεις Μακάλιστερ, είναι σωστές, ισορροπημένες. Μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι και δείχνουν την σωστή πορεία που ακολουθεί η Σερβία. Εγώ είμαι Σλοβένος, προέρχομαι από την πρώτη χώρα της τέος Γιουκοσλαβίας που έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι για τις επιλογές της Σερβίας. Έγιναν μεταρρυθμίσεις που ήσαν ταμπού πριν λίγο καιρό. Πρέπει όμως να συνεχιστεί η προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η Σερβία έχει πράγματι ανάγκη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για να μπορέσει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα την καταστήσουν μέλος της Ένωσης. Για ένα λεπτό ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η Σερβία έδειξε ότι θέλει να εμπλακεί πλήρω στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και να ενοποιήσει ευθέω και ρητά τις αναγκαίες μεταρρυθμίσει για να συνεχίσει να αλλάζει και να προσεγγίζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι διαπραγματεύσει σίγουρα δίνουν θετικά αποτελέσματα. Φερρυπίν, μια σειρά θετικών βημάτων στην, στην ε, διευκόλυνση των σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο και τις ε, γενικότερες δράσεις ε, ασφαλών, ασφαλές των σχέσεων με τη γειτονιά της αλλά και την ενίσχυση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σερβία είναι μια βαλκανική χώρα αλλά στρατηγική σημασία. Είναι προφανής λοιπόν η ανάγκη να ευθυγραμμίζει την εξωτερική της πολιτική, την πολιτική ασφάλεια με αυτή της Ένωσης. Η προσέγγιση, η ευθυγράμμιση των θέσεων της Σερβίας με της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασικό στοιχείο για την ευρωπαϊκή προοπτική και εύχομαι η κυβέρνηση του Βελγαδίου να κάνει τις αναγκαίες ε, και θαραλές επιλογές για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς για 1,5 λεπτό. Χαιρετίζω τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σερβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει όμως να δηλώσω ότι θα προτιμούσα να έχει δοθεί το δικαίωμα στους πολίτες της σερβίας να έχουν αποφασίσει με δημοψήφισμα για τη διαπραγμάτευση σχετικά με τη μελλοντική τους ένταξη στην ευρωπαϊκή ένωση. η ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της σερβίας και έχει συνάψει από το 2010 χιλιάδες δέκα συμφωνίες συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας πρέπει ορισμένα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης να μην θέτουν εμπόδια στον ευρωπαϊκό δρόμο της σερβίας και να συμφωνήσουν να ανοίξουν για διαπραγμάτευση και νέα κεφάλαια. ταυτόχρονα οι σερβικές αρχές οφείλουν να εντείνουν τη δράση τους για το χτύπημα της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. βεβαίως η επαρκής εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων καταδεικνύει ότι η σερβία υλοποιεί τις δεσμεύσεις της στον τομέα του κράτου δικαίου τη δημόσια διοίκηση και τη οικονομική διακυβέρνηση. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αποφάσισα να λάβω το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye, γιατί έχω μία ερώτηση ιδίω προ τον κύριο Πλένκοβιτς Μιλήσαμε στο σύντομο διάλειμμα σχετικά με την τροπολογία σας εξηγήσατε και τώρα τα θέματα ε, των αρμοδιοτήτων, αλλά θα ήθελα κάποιες ε, περισσότερες πληροφορίες. Ο νόμος ε, τον οποίο θέλαμε να καταργήσουμε με αυτή την τροπολογία ήδη από το 2003 είχε γίνει και το δέχτηκε και η Επιτροπή και η διεθνή Κοινότητα. Και η υπόθεση Μπέλγο αυτό κατατάσσεται και ε, ε, είχε δοθεί πλήρης τεχνική βοήθεια και νομική βοήθεια σύμφωνα με αυτόν τον νόμο στους βασικούς μάρτυρες και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί ε, θέλετε να το καταργήσετε. Νομίζω ότι είναι γενικότερη αρμοδιότητα και όχι μόνο για τη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Είχατε μόνο ένα λεπτό. Κύριε Πλένκοβιτς, θέλετε να απαντήσετε σε αυτό το σημείο και μόνο για 30 λεπτά έχετε το λόγο. Αγαπητή κυρία Λούνατσετς, εν μέρη βλέπω ότι έχετε πληροφορηθεί για το θέμα αυτό. Προτείνω να συζητήσουμε διμερώς το θέμα αυτό γιατί έχουμε μόνο 23 δευτερόλεπτα που μου έχουν μείνει. Το ότι ο νόμος είχε περάσει το 2003 δεν σημαίνει ότι υλοποιήθηκε μέχρι το 2010 και επί τη ευκαιρία η Κροατία έχει θεσπίσει ένα νόμο που ακυρώνει όλες τις νομικές πράξεις βάσει αυτού του νόμου μέχρι το 2011. Άρα είναι μεροληπτική η ενημέρωση που έχετε και έχετε το κατά νου μέχρι την ψηφοφορία αύριο. Τελευταία παρέμβαση, ο κύριος Κοστέλο. Ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει ξεκινήσει μια μακρά διαδικασία η χώρα αυτή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σημασία λοιπόν η αναφορά την οποία έκανε ο συνάδελφος Μακάλιστερ με την οποία συμφωνώ μαζί του. Είναι ιδιαίτερα ισορροπημένη, δεκτική και συμφωνούμε όλοι οι σκιώδεις εισηγητές τίθεται όμως το θέμα των, αγνοη... των αγνοουμένων. Είναι μια χένουσα πληγή αυτό στην ε, τέος Ιουκοσλαβία. 12.000 οικογένειες δεν γνωρίζουν τι έγιναν οι αγαπητοί, οι αγα... τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδιαίτερα σε περιοχές ε, γύρω από το Μόστα. Ε, έχει επίσης αναλάβει πρόσφατα στο παρελθόν και την προεδρία του ΟΑΣΕ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις στενές σχέσεις πολιτιστικές και θρησκευτικέ που έχει με τη Ρωσία. Ελπίζω να υπάρξει ε, διπλωματία και να σταματήσουν να πνέουν οι άνεμοι του πολέμου. Λοιπόν, δίδω το λόγο στον Επίτροπο Χάννα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, κύρια Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ευχαριστώ για την συζήτηση που δείχνει τη σημασία που δίνει η Ένωση στην ε, ενταξιακή στην διαδικασία και την υποστήριξη της διεύρυνσης στην περιοχή ιδίω. Καταγράφω ότι οι για την ε, νομοθεσία τη ουσία για το ρόλο των αρχών στις δίκες για θέματα για εγκλήματα, για εγκλήματα πολέμου. Τούτο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο μελλοντική συνεργασίας. Με την ίδια ευκαιρία θέλω να υπογραμμίσω ότι η αμερόληπτη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των, των εγκλήματων πολέμου που σέβονται τις διεθνεί προδιαγραφέ, είναι υψηλά στο, στις διαπραγματεύσεις Σερβία. Ιδίω ε, στο άρθρο 23 τη διαδικασία screening που αφορά το, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τι δικαστικέ αρχέ και όπου υπογραμμίζεται η ανάγκη αποτελεσματική και αμερόληπτη αντιμετώπιση των ε, εγκλημάτων πολέμου και ε, ίση αντιμετώπιση των ε, υπόπτων, αναλογικότητα και προστασία των θυμάτων. Όλες αυτές οι συστάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο τμήμα για το δικαστικό σώμα του προγράμματος δράσης που είναι απαραίτητο για την έναρξη του κεφαλαίου 26. Η Επιτροπή συνεργάζεται στην, ε, και εμπλέκεται ενεργά στην προετοιμασία του προγράμματος δράσης και παρακολουθεί τις δραστηριότητες της Σερβίας ε, στο πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και συγχαρητήρια και πάλι στον κύριο Μακάλιστερ και τους συναδέλφους του για την εξαιρετικά ισορροπημένη έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπο Χάν. Η κυρία Λουκασέβιτσα από το Συμβούλιο. Κυρίες και κύριοι, Επίτροπε, Πρόεδρε, κλείνοντας τη συζήτηση θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου πραγματικά για μια εξαιρετική δουλειά και γενικά για τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την πορεία της Σερβίας. Ο εισηγητή ο κ. Μακάλιστερ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν χρήσιμη η που προηγήθηκε. Η Σερβία τώρα πλέον μπορεί νομίζω να συνεχίσει τον δρόμο μπροστά της με περισσότερη ευκολία και άνεση. Πολλά βέβαια κεφάλαια δεν έχουν ανοίξει ακόμα, αλλά παρόλα αυτά η Σερβία δείχνει ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει την πρόοδο. Ε, και στα πλαίσια αυτά η, θα ανοίξει σύντομα το τρίτο κεφάλαιο. Εμείς βασιζόμαστε στις βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων. Λέγεται ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την προετοιμασία της χώρας ε, για ε, την ένταξη. Απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω πρόοδο σε επίπεδο κράτος δικαίου και σε επίπεδο σχέσεων με το κοσυφοπέδιο. Έτσι λοιπόν εμείς καλωσορίζουμε τον διάλογο υψηλού επίπεδου που ανακοινώθηκε ανάμεσα στις δύο χώρες στις αρχές Φεβρουαρίου. Πρέπει η όθηση αυτή να οδηγήσει τις δύο χώρες να καταλήξουν σε συμφωνίες και για τα υπόλοιπα θέματα. Εμείς θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ε, παρακολούθηση των βημάτων προόδου. πριν ξεκινήσουν οι επόμενες φάσεις της διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια που κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πείσει τη Σερβία να εντατικοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις είναι ιδιαίτερο θετική. Σας ευχαριστώ ε, για τη συμβολή σας στη συζήτηση. you, Ευχαριστώ. Κύριε Υφυπουργέ, ευχαριστώ και κύριε Μακάλιστερ για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε και ο κατάλογος των ομιλητών. Έχουμε πλέον λοιπόν τώρα την πρόταση ψηφίσματος. Α, θα ψηφίσουμε αύριο για αυτήν.